Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ για να ε, σας πω που βρισκόμαστε σε σχέση με ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και που τα συζητήσαμε και το καλοκαίρι. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρο, σήμερα το πρωί εγκρίναμε ένα σύνολο πακέτων ε, για τις ροέ ΗΠΑ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση εμπιστοσύνη, επί τη βάση της ομάδας εργασίας ad hoc και συμπεριλαμβάνει επίσης τα θέματα TFTP, TFTS και PNR. Θα επικεντρωθώ σε αυτά τα τρία λοιπόν αναφέροντας ότι ε, υπάρχει και το θέμα του ασφαλούς ε, ε, λιμένα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο και θα το αφήσω στην συνάδελφο να σας μιλήσει γι' αυτό. Για τα δεδομένα TFTP είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει πριν από τη σημερινή συζήτηση, από τότε που άρχισε το θέμα του NSA Εγκρίναμε αυτή την αξιολόγηση όπως αναφέρθηκε και στην ε, συμφωνία τρία χρόνια μετά την ε, έναρξη ισχύω. Δεν είναι αναθεώρηση Σκοπό έχει να αξιολογήσει την αξία των δεδομένων αυτών, ε, των δεδομένων που διατηρούνται για πολλά χρόνια και των ε, ωφελών που έχει κάτι τέτοιο για την αντιμετώπιση των ε, δραστηριοτήτων τρομοκρατίας. Η έκθεση παρουσιάζει διάφορους τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα TFTP μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη και αυτές οι επεξηγήσεις συνοδεύονται από πραγματικά περιστατικά. Ε, κάναμε πολύ σκληρή δουλειά για να εντοπίσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ε, που αποδεικνύουν ακριβώς ε, ότι τα δεδομένα TFTP βοηθούν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Είχαμε απόρριτες συναντήσεις με τα κράτη-μέλη και με τη Europol που συμμετείχε στην έκθεση. Πάνω από χίλιες εκθέσεις TFTP έγιναν ε, και ήρθαμε σε επαφή με πολλούς ερευνητές TFTP. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση και τα οποία μπορείτε να, να εξετάσετε πιο προσεκτικά μετά τη συνεδρίαση. Ε, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά ε, για ε, την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών, για παράδειγμα στη Συρία και δείχνει ακριβώς τη σημασία των δεδομένων TFTP για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση των τρομοκρατών και των δικτύων υποστήριξής του σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως επίσης και νέα δίκτυα υποστήριξης. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να υπάρξουν νέες αποδείξεις και για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε πληροφορίες από άλλες πηγές. Όσον αφορά την ηλικία των δεδομένων αυτών είναι προφανές ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την ε, αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Όταν συμφωνήσαμε για το θέμα των δεδομένων TFTP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ένα πλαίσιο για τη χρήση των δεδομένων αυτών σε ευρωπαϊκό έδαφος ε, και την δημιουργία ενό συστήματο ε, ισοδύναμου του TFTP και το σύστημα που έχετε μπροστά σα είναι αποτέλεσμα μιας διεξοδικής διαδικασίας αξιολόγησης ενό συστήματος που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τι απαιτήσει ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει μια εξωτερική μελέτη, έχουν συμπεριληφθεί πολλοί ανεξάρτητοι φορείς από το Ευρωπόλ, ε, από διάφορους παρόχους υπηρεσιών, ε, δεδομένων TFTP. Είδαμε διάφορες δυνατότητες για να υπάρξει μια συζήτηση. Το κάναμε αυτό το 2011 και παρουσίασα τότε τα αποτελέσματα. Δεν υπήρξαν σαφείς ε, ενδείξεις από εσά για το πώς θα θέλατε να προχωρήσουμε. Κάποια κράτη-μέλη είπαν ότι η ε, άγκληση δεδομένων ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ενδεχομένω μια πιθανότητα. Το λάβαμε υπόψη στην αξιολόγηση, αλλά δεν είχαμε μακρά συζήτηση ούτε στο Συμβούλιο. Είδαμε τι διάφορε επιλογέ βάσει των αρχών ε, τη στρατηγική διαχείριση των πληροφοριών, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και σχέση κόστου αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά το καθεστώ διατήρηση και άντληση δεδομένων, δεδομένων τονίστηκε από εσά ότι ήταν ένα τρόπο ε, να υποστηριχθεί το πλαίσιο τη άδληση δεδομένων στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ε, σε αυτή την περίπτωση θα μετακινείται το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως αυτό δεν θα σήμαινε επιπλέον ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε θα εξασφάλιζε καλύτερη προστασία των δεδομένων. Η Προστασία στα ε, πρόσβαση στα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να έχουμε μια στεναρή ε, προστασία δεδομένων. Ε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν έρευνες αυτή τη στιγμή, ε, έρευνες για τα δεδομένα αυτά. Πρέπει να υπάρξει μια ξεχωριστή βάση δεδομένων και αυτό βέβαια θα σήμαινε σημαντικό κόστος, πόρους και επίσης πολύ περισσότερη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμόρφωση με τις ρήτρες προστασίας των, προστασίας των δεδομένων. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρξει πράγματι μια διαφορετική βάση δεδομένων, μια άλλη βάση δεδομένων αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το ανεξάρτητο σύστημα τώρα, είδαμε διάφορες ε, πιθανότητες για να διευκρίνουμε το σύστημα, για παράδειγμα διαφορετικές μεθόδους πληρωμών και συγκεκριμένους παρόχους ε, υπηρεσιών. Γιατί αν υπάρξει ένα νέο σύστημα, τα μελη -μέλη, πολλά κράτη-μέλη θα το επιθυμούσαν αυτό παρά το γεγονό ότι η προθυμία για τέτοιου είδου σύστημα είναι πολύ περιορισμένη στο Συμβούλιο. Όμως θα μπορούσε να, διευρύνει, να διεπεκτείνει τι δυνατότητές μας για την αντιδρομοκρατική δράση όμως είναι ένα πολύ απαιτητικό, ε, δαπανηρό ε, σύστημα και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο αυτό είναι αναλογικό με το στόχο μας. Επίσης αποκλείσαμε δύο μη ρεαλιστικές προσεγγίσεις, το πλήρες ε, κεντρικό σύστημα μόνο ευρωπαϊκό και ένα απολύτως αποκεντρωμένο το οποίο θα είναι υπό τη διαχείριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι μεικτό. Κάποιες αρμοδιότητες θα είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, λεπτομέρειες θα δείτε και στην έκθεση. Θα μπορούσε τότε να εξοπλίσει με ένα ανεξάρτητο σύστημα ε, έρευνας την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπό το φως βέβαια πολύ συγκεκριμένων εξελίξεων, κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ δαπανηρό, χρονοβόρο και δύσκολο να, στη συντήρησή του. Και θα σήμαινε επίση και τη δημιουργία μιας τελείως καινούριας ε, βάσης δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβάλει τη σχετική πρόταση, θα τα αφήσουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να το συζητήσουν και να υποβάλουν τις συστάσεις τους ενδεχομένως για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ξέρω ότι καθυστερώ λιγάκι κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι πολλά στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στην ε, έκθεση και θέλω να είμαι ω το δυνατόν πιο διεξοδική. Μία κοινή επίσης αναθεώρηση θα έχουμε για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για το PNR το καλοκαίρι έγινε αυτό, εμπειρογνώμονες ε, έλεξαν κατά πόσο ε, το, Υπουργείο Εσωτερικών, ε, το σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών της Αμερικής συνάδει με τα δικά μας πρότυπα και είδαμε ότι όντως πράγματι η λειτουργία του ο φιλτράρει δεδομένα ε, για τις πτήσεις ε, και μόνο, δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα για άλλους λόγους ε, και η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, η διαχείρισή τους, η μεταφορά τους γίνεται μόνο επί συγκεκριμένων περιπτώσεων και έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν βέβαια περιθώρια βελτιώσεων όσον αφορά την εξέλιξη της συμφωνίας αυτής εννοώ για την ε, διαγραφή και την ε, αποπροσωποποίηση των δεδομένων, την διαγραφή τους από το σύστημα. Τώρα γίνεται μερικές ημέρες ε, μετά, όταν ενημερώνεται το σύστημα. Επίσης προχωρούμε ως προς τη χρήση της μεθόδου push and pull. Έχουμε μια καλύτερη ε, αξιολόγηση των δεδομένων, 0,13% ε, όλων των δεδομένων PNR ε, είναι αντικείμενο της μεθόδου, έχουν προκύψει από τη μέθοδο pool, η οποία λοιπόν χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Επίσης ζητούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αμοιβαιότητα και την αστυνομική συνεργασία, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους μηχανισμούς αποζημίωσης. Η έκθεση αναφέρει επίσης ε, ότι το Υπουργείο των Ηνωμένων Πολιτειών ε, προβλέπει κοινοποίηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός 48 ώρων από την πρόσβαση των δεδομένων ε, κάθε τρίμηνο αναθεωρούν τους κανόνες και τις ανάλυσεις ε, των στόχων ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση ή να αποφεύγεται αυτή. Επίσης ε, προτείνεται να επισπευτεί διαδικασία της διαδικασίας push μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εντάχει στις συζητήσεις ε, για το TFTP και την έκκλησή σας ε, για αναστολή της συμφωνίας. Επειδή έχουμε διαβάσει σχεισμούς ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόσβασης των Ηνωμένων Πολιτειών μη εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αρχίσει έρευνα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας και υπήρξαν πάρα πολλές επαφές, τηλεφωνικές, αλλά συνάντησα κιόλα, ε, και συζήτησα με τον David Cohen εδώ ε, στις Βρυξέλλες, αλλά και στη Washington την περασμένη εβδομάδα. Πήγα και στο Λευκό Οίκο, μίλησα και με τον ε, υπεύθυνο ασφαλείας του Προέδρου. Ο κύριος Κοέν λοιπόν γραπτός με διαβεβαίωσε ότι δεν ε, έχει υπάρξει παραβίαση από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών. Σας έχω αποστείλει και τις σχετικές επιστολές ε, για να ε, τις διαβάσετε και μόνοι σας. Μιλήσαμε για όλα τα στοιχεία. Δεν έχω λάβει κανένα αποδεκτικό στοιχείο ότι υπήρξε παραβίαση της συμφωνίας. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτε τέτοιο. Επίσης ήμασταν ε, σε πολύ στενή επαφή με τον ε, πάροχο υπηρεσιών, ε, τον εγκεκριμένο τη SWIFT και μας είπαν και εκείνοι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι, ενδείξεις παραβίασης της συμφωνίας. Θα έχουμε επίσης λεπτομερή εξέλιδαση του θέματος αυτού και στο μέλλον. Την άνοιξη θα γίνει νέα αναθεώρηση αποφάσισα να κλείσω τις διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις με όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις σας, ε, σας ανέφερα. Έστειλα και σχετική επιστολή που επίσης έχω συμπεριλάβει στο φάκελο. Η Υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης ε, εμπιστοσύνης, ε, ε, αύξηση της συμμετοχής τους στις διαβουλεύσεις και στις διαδικασίες. Θα το δείτε άλλωστε και στο, στις επιστολές. Ε, εγώ ακόμη έχω, είμαι σοκαρισμένη από όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έκανε ο Σνόουντεν σε σχέση με τις ε, διάφορες, ε, με, με τους τρόπους με τους οποίους οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Ευρωπαίους και συνεπώς πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουν οι σχέσεις μας όπως ήταν πριν. Το συζητήσαμε πολλές φορές και στην, και στην ανακοίνωση που σήμερα εγκρίναμε μαζί με την Επίτροπο Ρέντινγκ και την ύπατη εκπρόσωπο Κάθριν Άστον. Έχουμε μια ιδέα των μέτρων αυτών. Μιλάμε για, την Ευρω... για τη μεταρρύθμιση των... της προστασίας των δεδομένων. Μιλάμε για ελπίδες ολοκλήρωσης της συμφωνίας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες μέχρι την Άνοιξη ή το καλοκαίρι και επίσης η Αντιπρόεδρος Έντινγκ θα μιλήσει για την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων του ασφαλούς λιμένα. Θα συζητήσουμε επίσης ε, το ενδεχόμενο περαιτέρω ε, συζητήσεων για το θέμα αυτό και επίσης με το Αμερικανικό Κογκρέσο συζητούμε συνεχώς ε, και προσπαθούμε να δούμε πώς οι μεταρρυθμίσεις που συζητιούνται στο Κογκρέσο και στη Γερουσία μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να είναι καλύτεροι ε, οι κανόνες, να υπάρχει ένας περιορισμός του τι μπορεί να κάνει η NSA, μεγαλύτερη παρακολούθηση, περισσότερη λογοδοσία, αλλά θα μπορούσαμε και εμείς ως Ευρωπαίοι να έχουμε μια καλύτερη ιδέα του τι συμβαίνει, και άλλες τρίτες χώρες βέβαια γιατί πάρα πολλοί πολίτες ε, Αμερικανοί και εκείνοι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από όλες αυτές τις αποκαλύψεις ε, παρακολούθησης. Αυτά. Εντάχει κυρία Πρόεδρε, σίγουρα θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, ευχαρίστως να προσπαθήσω να τις απαντήσω ε, όσο λεπτομερέστερα μπορώ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μπορεί να μην έχετε διαβάσει όλα τα έγγραφα, αλλά ευχαρίστως να απαντήσω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 Λοιπόν, ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας παρουσιάσατε τα γεγονότα. Είπατε πως υπάρχει χώρος ε, για βελτιώσεις. Τι εννοείται βελτιώσεις. Είναι αυτό το οποίο συμφωνήσαμε ως συνθήκη γενικά σε καλές γραμμές εντάξει και κάτι ψηλολεπτομέρειες δεν πάνε καλά ή θα ή είναι του τύπου ε, ενός μεγάλου κενού στην προστασία των δεδομένων. τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή είναι σοβαρά τα προβλήματα ή λιγότερο σοβαρά. Θα μείνω σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε μερικές ερωτήσεις ακόμα. Ο κύριος Μωραές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κίνγκα. Ναι, συμφωνώ. Πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τις ποιοτικές βελτιώσεις και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι δύσκολο γιατί δεν είχαμε ευκαιρία να δούμε την ανακοίνωση εις βάθος. Αλλά νομίζω πως ε, κάνατε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε μαζί μας ε, και κάνατε τα πάντα εγκαίρως. Επίσης, στο μέλλον η διαδικασία διαβούλευσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια νομίζω και αυτό είναι θετικό. Από αυτά που είδαμε λοιπόν από την ανακοίνωση, το μέλλον είναι λαμπρό. Ο δε κύριος Βος ρώτησε σωστά ποια θα είναι η ποιότητα αυτών των βελτιώσεων. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να τα αξιολογήσουμε αυτά. Κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε είναι το πού θα κλείσει αυτό το θέμα. Μιλήσατε για το ότι δεν ετέθη ζήτημα παραβίασης της πρόσβασης των δεδομένων. Πρέπει να δούμε το ψήφισμα λοιπόν του Οκτωβρίου και να σας υπενθυμίσω και πάλι πως όταν μιλάμε για προσωρινή αναστολή της συμφωνίας TFTP υπήρχαν τρεις όροι εδώ πέρα που έχουν εκπληρωθεί. Το βασικό είναι αυτά τα οποία ακούστηκαν για παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα από την NSA. Μετά είχαμε την επιστολή σας στις 26 Νοεμβρίου στον Υπουργό, τον κύριο Κοέν. Είπατε πως ε, μαζί με τις πληροφορίες που λάβατε συμπεραίνεται πως οι ΙΠΑ είχαν δράσει με τρόπο αντίθετο με τη συμφωνία SWIFT. Ε, δεν είχαν δράσει με τη συμφωνία, και πως ε, η συμφωνία ήταν και παραμένει σεβαστή. Από ό,τι καταλάβαμε, το αντικείμενο ήταν μόνο το εάν είχε χακαριστεί το σύστημα SWIFT και αν είχε πρόσβαση η NSA ή κάποιος άλλος. Ε, αυτό το οποίο είπαμε εμείς στο ψήφισμά μας όμως προς Συμβούλιο Κομισιόν και είπα ήταν πως υπήρχε πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα με τρόπο άλλο εκτός του SWIFT. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως οι βουλευτές δεν μιλούσαν για άλλους άλλους νόμιμους τρόπους πρόσβασης. Οπότε ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα. Και πρέπει να πω πως αντιλαμβάνω πως δεν έχετε δει ακόμα επαρκώς αυτές τις κατηγορίες. Πριν κλείσει λοιπόν το θέμα χρειάζεται μία απάντηση. Το ζήτημα λοιπόν είναι μεγάλο ακόμα και δεν θεωρώ πως έχουμε κάνει τη δουλειά μας μέχρι να λάβουμε μια απάντηση σχετικά. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φως. Είναι ζήτημα πλέον ανάλυσης των σχέσεων μας και δεν μπορούμε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό πριν έχουμε, έχουμε μια σαφή απάντηση. Σας ευχαριστώ Κλοντ. Σοφή Νετφέλντ. Με ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ήρθε η Επίτροπος για να παρουσιάσει τα έγγραφα αυτά και θα τα διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ όμως με τους δύο προλαλήσαντες. Ο Κλόντ είπε πως το κεφάλαιο δεν μπορεί να κλείσει. Μιλώντας με την ίδια παρομοίωση, θυμάμαι εγώ τα παιδικά παραμυθάκια που διάβαζα Όταν λοιπόν μιλάμε για έρευνα όπου η Κομισιόν ρωτάει την NSA μπήκατε στο σύστημά μας παράνομα και η NSA λέει μα όχι εμείς. Ε, αυτό είναι κόκκινο σκουφίτσα έτσι. Έφαγες τη γιαγιά μου. Όχι απαντάει ο Λύκος. Ε, συγγνώμη δεν είναι έρευνα αυτό. Έτσι. Το Swiss είπε πως έκανε το δικό της έλεγχο. Ωραία, ε, εμείς πώς το επαληθεύουμε. Γιατί δεν έγινε, όπως ζητήσαμε, επί τόπου μία έρευνα τεχνολογική ε, η οποία θα η, με μεθόδους της σήμανσης η οποία θα είχε οριστικά αποτελέσματα. Αλλιώς ναι, ρωτάμε την NSA και ορκίζεται στην προσκοπική της τιμή. Αλλά αυτό δεν είναι έρευνα. Δηλαδή συγκινητικά αυτά που μας λέτε, αλλά δεν μας πείθουν. Οπότε, αν μιλάτε πραγματικά για μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ε, δεν είναι αυτά. Μετά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την αναστολή της συμφωνίας ε, SWIFT ή TFTP και η απάντηση της Κομισιόν είναι σας αγνοούμε και ανταυτού προτείνουμε μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία TFTP. Και αυτό δεν ε, μας ε, εμπνέει η εμπιστοσύνη. Επίσης ζητήσαμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα άντλησης δεδομένων, όχι ένα ευρωπαϊκό σύστημα TFTP. Μετά, πού ήταν η περιγραφή. Ο λόγος για τον οποίο απορρίπτεται ένα σύστημα εξαγωγής των δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος γιατί θεωρείται πως οι Αμερικανοί θα μπορούν απευθείας από την βάση δεδομένων να κάνουν την εξαγωγή. Όχι. Εμείς θέλουμε να μας ζητάνε συγκεκριμένα δεδομένα και οι δικοί μας δικοί να κάνουν την εξαγωγή, όχι πρόσβαση των Αμερικάνων. Και ενδιαφέρον, επίσης, αυτό το οποίο λέτε, ότι η SWIFT δεν μπορούσε να το κάνει αυτό από μόνη της, γιατί η βάση δεδομένων που έχει δεν επιτρέπει αναζητήσεις με βάση προσωπικά δεδομένα. Μα ε, αυτή δεν είναι η βάση της συμφωνίας. Αν δεν μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα δεδομένα, τότε εξορισμού αυτό το οποίο λέτε είναι πως τεχνολογικά μπορούν να δώσουν δεδομένα μόνο μαζικά. Οπότε η συμφωνία ε, αυτομάτως είναι άκυρη, έτσι, γιατί το νόημα ήταν να μειωθούν τα δεδομένα που μεταφέρονται. Οπότε ε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Διαβάζω προσεκτικά τα δεδομένα. Ειλικρινά δεν με καθησυχάζουν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη είναι πλέον θέμα κατεπήγων. Όχι με τη ΣΥΠΑ, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και Κομισιών και μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων μεταξύ των οποίων και εκτελεστικά όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήλπιζα να διαβάσω τα έγγραφα και να με καθυσυχάσουν, αλλά όπως λέει και ο Κλοντ δεν μπορεί να κλείσει έτσι αυτό το κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ κύριε Κέρκοπ. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ ελάχιστα με την προηγούμενη λίτρα. Μα θα ανησυχούσα, λέει η κυρία Ινετφέλντ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως ε, εγώ ε, εκτιμώ το έργο της Κομισιόν, εξάλλου είναι ευθύνη της Κομισιόν και όχι του Κοινοβουλίου θα έλεγα εγώ και η Κομισιόν κινήθηκε εξαιρετικά γρήγορα και συγχαίρω την κυρία Μάστο και νομίζω πως οφείλουμε να ε, δεχτούμε θετικά την πρωτοβουλία της Κομισιόν για επανεξέταση των συμφωνίων, κάτι το οποίο θεωρώ, εκτός βεβαίως αν κανείς είναι καχύποπτος για τα πάντα, αρκεί για να καθησυχάσει α, ε, λογικούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ε, επανακτήσουμε την ε, εμπιστοσύνη και βεβαίως θα το περιμένουν αυτό στην συνάδελφοι. Η ΕΠΑ ΕΕ είναι πάρα πολύ σημαντικός σύμμαχος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Είχαμε και πρόσφατες εμπειρίες και πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην διακινδυνεύσει η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι βασικό για εμένα και θεωρώ πως πρέπει να διαχωρίσουμε το ζήτημα της συλλογή πληροφοριών και τις σχετικές υπηρεσίες με τις καθημερινές αστυνομικές επιχειρήσεις και συνεργασία που έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε υπέρ της ε, δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης ε, της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και να πω και εγώ λίγο κάτι, μια που είμαι εδώ πέρα αρκετά χρόνια, που προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικών επιβατών. Δηλαδή, αν είμαστε λογικοί, όσοι ε, ανησυχούν για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ θα έπρεπε να θέλουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, δεδομένων αεροπορικών επιβατών στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ πέρα, ε, λίγο περίεργη. Επίσης, θα ήθελα να πω πως Ξέρετε, οι συμφωνίες είναι όλες σημαντικές αυτές για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Επίσης, εμένα με καθησυχάζει το ότι η Europol θεωρεί πως οι συμφωνίες αυτές αυξάνουν την ασφάλεια και ε, η παρακολούθηση της χρηματοδότησης νομίζω έχει αποδειχθεί ε, πάρα πολύ σημαντική όπως αποδείχθηκε και με την υπόθεση Breivik και με τις ε, βομβιστικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου. Οπότε το Κοινοβούλιο μιλάει για δικλείδες ασφαλείας, αλλά δεν θέλει να κάνει κάτι για να δώσει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τους πολίτες της Ένωσης. Εγώ ελπίζω να προωθήσουμε θέματα της αρμοδιότητάς μου, αλλά εν μεταξύ θεωρώ πως πρέπει να συγχαρούμε και πάλι την Κομισιόν. Είναι, όπως είπα, ευθύνη πρωτίστως της Κομισιόν και η Κομισιόν μου φαίνεται πως ε, έχει σωστά εξασκήσει τα καθήκοντά της και πρέπει να την επενέσουμε. Σας ευχαριστώ, θα παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Για να δώσω τον λόγο σε όλους. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάλμστρομ για την παρουσίασή της. Κατρεχάς, για την σας να πω ότι πολλά σημεία βλέπω σε ολόκληρο το πακέτο της ανακοίνωσης ε, που είναι πολύ χρήσιμα για τις ε, μενόμενες διαπραγματεύσεις ε, σε σχέση με ολόκληρο το θέμα ε, της ε, ροής ε, δεδομένων και της προστασίας δεδομένων και νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα σημεία αναφερόμενοι στον τεράστιο όγκο διασυνο... διατλαντικής μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων. Βέβαια, στο πλαίσιο των υπολείπων ε, συμφωνιών επιβολή του νόμου θα ήταν σημαντικό να έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία ε, προστασίας δεδομένων. Ε, κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε τέτοιου είδους συμφωνίες χρειαζόμαστε μια συμφωνία ευρύτερη και μας, ε, ε, μας ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αλλάξει η νομική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών για την κάλυψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων πολιτών που δεν αναφέρονται για την ώρα όταν μιλάμε για την αποζημίωση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάντοτε στο πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων και πρέπει να επιμείνουμε γι' αυτό. Αλλά για να επιμείνουμε Νομίζω ότι πολύ σοφή απόφαση αυτού του Κοινοβουλίου ήταν να πει ότι αν δεν υπάρχει κίνηση και δεν υπάρχει ε, κίνηση, αν υπάρχει παρέκκληση ε, όλων των ρητρών ασφαλείας, των δικλείδων ασφαλείας που έχουμε, πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες και οι, οι συνέπειες αυτές ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την αναστολή της συμφωνίας TFTP. Δεν θέλω να ξαναμπούμε στη συζήτηση αυτή, αλλά το ζητήσαμε και το αγνοήσατε παντελώ. Είναι ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα αυτό. Είναι ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα, γιατί αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υποβάλλει αιτήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς τα αγνοεί, ε, δεν μπορούμε να το δεχθούμε κάτι τέτοιο και το αναφέραμε στο ψήφισμα το οποίο υπερψήφισε η πλειοψηφία, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την έγκριση των ε, μελλοντικών ε, διεθνών συμφωνιών, γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι συμφωνίε, ούτε μπορούμε να θέσουμε ένα όριο ε, πουθενά, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια αγνοεί τα αιτήματά μα για το TFTS και το, το, το σύστημα TFTS, Αναγνωρίζω το γεγονός ότι το σύστημα αυτό μπορεί να μην είναι τόσο πολύ αναλογικό, αλλά όπως είπε και η κυρία Ινιτφελ, ζητήσαμε μία μέθοδο άντλησης να έχουμε εξατομικευμένα στοιχεία τα οποία θα αντληθούν να υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή δεδομένων για μια συγκεκριμένη υποψία, για ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Αυτό είναι η ίδια η φύση του ε, κανόνα δικαίου που έχουμε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση των δεδομένων αυτών, υπό καμία άλλη έννοια, εκτός αν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη υποψία και σε συγκεκριμένο κίνδυνο. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω. Διάβασα στο Huffington Post ότι γίνονται πλέον ε, ε, καταγραφές όλων των προσβάσεων σε πορνογραφικά sites ε, γιατί θεωρείται ότι μπορεί με τέτοιο τρόπο να ριζοσπαστικοποιούνται Μπορεί κάποιο να καταλάβει έτσι τι σεξουαλικέ κλήσει κάποιων άλλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμω είναι εντελώ απαράδεκτο. Είναι κάτι που αποδυναμώνει, υπονομεύει το κράτο δικαίου μα και δεν ακούω τίποτε, δεν διαβάζω τίποτε σαν ανακοινώσει σα που να το καταδικάζει αυτό. Η επιτήρηση, η αποπτία έχει αποτύχει. Πρέπει εμείς να ε, το σταματήσουμε αυτό πρέπει να είναι διαφορετική η, αντιμετώπιση, η διαφορετική αντιμετώπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο, στο, στο, στο σύστημα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις ε, σε σερβερς ε, από ε, ξένες αρχές είτε μέσω εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, να πω πως έχουμε άλλους 7 ομιλητές. Έχουμε άλλους 7 ομιλητές εδώ πέρα, οπότε σας παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι. Ε, δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά ε, να είστε σας παρακαλώ σύντομοι. Για να μιλήσουν όλοι. Κατόπιν η Κυρία Έρνστ, σας ευχαριστώ. Επιτρέψατε μου, κυρία Μάνστρομ. Το έγγραφο αυτό μου θυμίζει τα έγγραφα της ε, λαοκρατικής δημοκρατίας Γερμανίας που μιλούσαν πάντα για την αδιάσπαστη φιλία με τη Σοβιετική Ένωση. Η ίδια λέξη συνέχεια. Έτσι που έφτανε να, να γίνεται γελία. Έτσι μου, αυτό μου θυμίζει. Και έχω πάθει αλλεργία απέναντι σε αυτή την αδιάσπαστη ενότητα από την νεότητά μου, το καταλαβαίνετε. Οπότε με, με, με συγχωρείτε αν είμαι λίγο κοινική, αλλά σοβαρά τώρα, δηλαδή αυτά τα οποία γράφετε εδώ πέρα στην έκθεση δεν επαρκούν με καμία δύναμη. Να πω κάποια πράγματα. Λέτε τι ωραία πράγματα έχετε επιτύχει. Ας δούμε λίγο λοιπόν τι απαριθμείτε στο παράρτημα θα διαπιστώσετε εκεί πως αναφέρονται γεγονότα τα οποία δεν έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Και δεν υπάρχουν γεγονότα των τελευταίων ε, ετών. Έτσι, τρομοκρατικά. Ε, αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια απόδειξη ότι το SWIFT πραγματικά συνεισέφερε κάπως. Δηλαδή Εάν μέσω των δεδομένων του SWIFT υπήρχε κάτι το οποίο έχει εμποδιστεί, θα είχε κάποια συνεισφορά. Τότε πραγματικά θα ήταν απολύτως απαραίτητο να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Τίποτα δεν υπάρχει, ούτε τεχνολογικά μας εξηγείται πώς λειτουργεί, ούτε με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Έτσι, τα είπανε και οι συνάδελφοι, δεν είναι πρόοδος. Μετά, ε, αναστολή της συμφωνίας. Είπατε πως έχετε γραπτή διαβεβαίωση, ερχόμαστε πάλι δηλαδή στην φιλία με τη Σοβιτική Ένωση, ότι δεν, ε, δεν βρήκαν δεδομένα. Μα με τι αποδείξεις. Τι αποδείξεις έχετε για το ότι όντως συμβαίνει αυτό. δηλαδή η διαβεβαίωση η αρκεί, να σας διαβεβαιώσω κι εγώ, έτσι. Συγκεκριμένα ποια δεδομένα έχετε, ποια υλικά, ποιες αποδείξεις για να επιβεβαιώσετε αυτό το πράγμα ε, κατόπιν. ερεύνησε κάποιος ε, το τι έγινε, το πώς κατέληξε η SWIFT, η NSA συγχωρείτε να μπει στο SWIFT. Το ερεύνησε κανείς. Πρακτικά επαλήθευσε κανείς αν ισχύει αυτή η κατηγορία. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη ΣΥΠΑ, οποιοδήποτε. τι συγκεκριμένα αποτελέσματα υπάρχουν. Όχι γραπτές διαβεβαιώσεις, συγκεκριμένα πράγματα. Πριν μιλήσουμε δε για ευρωπαϊκό SWIFT ή SWIFT ε, Lite ή με την ε, φιλική χορηγία της NSA, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να ξεχαρίσουμε τουλάχιστον αυτό το ζήτημα λέτε πως έκλεισε αυτό το θέμα και εντάξει όλα καλά, δεν χρειάζεται έρευνα, δεν χρειάζεται να αναστείλουμε τη συμφωνία. Τίποτα δεν έχετε ως απόδειξη. Και για την υπόθεση του PNR. Λέτε πως στηρίσατε τις συνθήκες. Πάλι, αποδείξεις, αποδείξεις. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου δηλαδή. Πρέπει κάποια στιγμή να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένα γεγονότα. Με την άγνοια αυτή δηλαδή της πραγματικής κατάστασης, ε, ε, κοινοβούλιο και κομισιόν και συμβούλιο γινόμαστε καταγέλαστοι από τους πολίτες. Τους πολίτες θα πάνε να ψηφίσουν έτσι. Τι θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. δικαιώματα εδώ πέρα παραβιάζονται χωρίς καμία αναστολή και μας λέτε ε, πως εντάξει το δεχόμαστε και δηλαδή το, το απορρίπτουμε ως απαράδεκτο αυτό το έγγραφο εδώ πέρα που μας έχετε δώσει. Σας ευχαριστώ Κορνίλια. Η κυρία Σίπελ. Do my best. Aber ich muss... Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορώ καν να το διαβάσω όλο αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί. Έχει πληγεί η εμπιστοσύνη προς τη ΣΥΠΑ, πρέπει να ανακτηθεί, αλλά ε, αυτό δεν γίνεται με τις υποσχέσεις των ΗΠΑ. Έτσι, ενοχλούμε γιατί ένα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, που λέτε δεν είναι καν δική σας υπόθεση, δηλαδή προστασία δεδομένων. Και από την άλλη, και το ευρωπαϊκό πακέτο και η συμφωνία ομπρέλα με τις ΗΠΑ με τα α, συμβάντα τα γεγονότα δεν έχουν απολύτως ουδεμία σχέση. Το συζητάμε πάνω από δύο χρόνια. Ναι εντάξει ωραία προστασία δεδομένων αλλά δεν έχει απολύτως ουδεμία σχέση με ε, αυτά τα οποία έκανε η NSA. Αυτό από μόνο του δεν είναι δυνατόν να αποτελεί μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Εγώ θέλω ξεκάθαρους κανόνες, ξεκάθαρες διαδικασίες για τις μυστικές υπηρεσίες. Και λέω μυστικές υπηρεσίες γιατί δεν είναι μόνο η NSA οπωσδήποτε, αλλά ιδιαίτερω αυτή. Μετά για το SWIFT. Ένα σημείο το οποίο αναφέρεται και λέτε δεν μπορούμε να έχουμε εξαγωγή των δεδομένων στο ευρωπαϊκό έδαφος είναι το κόστος. Το κόστος. Σοβαρά. Όλα τα υπόλοιπα αντιτρομοκρατικά χρηματοδοτούνται. Προσπαθήσαμε να το βγάλουμε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ένα συνάλφο μάταια. 50 εκατομμύρια για το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σίγουρη πως θα έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα ελέγχου των συνόρων επίσης δωρεάν. Όλα αυτά κοστίζουν λεφτά, έτσι παρά την κρίση, κανένα πρόβλημα δεν έχετε, μόνο για τα δεδομένα του SWIFT ξαφνικά δεν υπάρχει μία. Και μετά είπατε και ελπίζω να σας άκουσα σωστά, πως δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα δεδομένα τα οποία θα, θα θέλαμε για την προστασία των δεδομένων τι προδιαγραφέ τι οποίε θα θέλαμε. Ε, δηλαδή, άμα δεν μπορούμε κι εμεί να τηρούμε τι δικέ μα προδιαγραφέ, τι, τι να πάμε να πούμε στου Αμερικάνου. Και τρίτον, λέτε δεν ε, θα χρησιμεύε σε τίποτα παραπάνω. Μα και εδώ πέρα ενοχλούμε. Μα ο σκοπό τη εξαγωγή των δεδομένων δεν είναι πλέον να πηγαίνουν χίδιν χοντρικά τα δεδομένα στις ΗΠΑ, αλλά εμείς να τα φιλτράρουμε και να τα δώσουμε σε τρίτη χώρα μόνο τα συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο αίτημα. Εγώ θεωρώ πως αυτό από μόνο του είναι προστιθέμενη αξία. Ενοχλούμε πραγματικά. Δεν νομίζω λοιπόν να μπορέσω να το ξεπεράσω έτσι εύκολα και για το ευρωαμερικανικό PNR νομίζω χρειάζεται λίγο περισσότερη ε, εμβάθυνση γιατί με αυτά που μας είπατε δεν αλλάζει τίποτα. Σας ευχαριστώ κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ. Μου κάνει εντύπωση που η κυρία Μάλμπστρομ, χαίρομαι βεβαίω ε, που είναι εδώ μαζί μας, που μπόρεσε να γράψει ε, στο στο Υπουργείο Οικονομικών ε, χωρίς να έρθει σε επαφή μαζί μας δεδομένου ότι εμείς ζητήσαμε την αναστολή της συμφωνίας και θα ήταν ίσως και από τακτικής απόψεως καλύτερο να ε, έρθει σε εμά και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό πριν από τη διαδικασία αποστολής επιστολών στο Υπουργείο Οικονομικών ε, που το έκανε χθε αυτό βέβαια. Τι να σας πω, εμένα, εγώ συνήθως δεν είμαι επικριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό Θα μπορούσατε να το γράψετε σήμερα, αφού ερχόσασταν εδώ. Πριν από μερικού μήνε το είχα ξαναρωτήσει. Πότε δεν κατάλαβα εγώ την επιστολή τη 18 η Σεπτεμβρίου του κυρίου Κοέν. Αλλά τέλος πάντων μου φαίνεται ότι γράφει αυτή η επιστολή όσο καταλαβαίνω ότι το TFTP δεν είναι πλέον η μοναδική πρόσφαση ε, στα ε, δεδομένα γιατί λέει ότι αφορά για παράδειγμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έρευνες που έχουν να κάνουν με, εγκληματο, με, με εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματίες. Μέχρι, μέχρι εκεί καταλαβαίνω. Δεν διάβασα την έκθεση βέβαια, δεν πρόλαβα, αλλά καλύπτεται στην έκθεση ότι υπάρχουν άλλες δύο άντλησης δεδομένων SWIFT. Γιατί μετά λέει, ότι ο κύριος, μετά λέει ο κύριος Κοέν λέει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το GFGP για να πάρει δεδομένα SWIFT τα οποία δεν μπορεί να τα λάβει από άλλες πηγές πριν από δύο μήνες το είπα, εγώ αφελώς δεν γνώριζα ότι είναι ε, η τελευταία μας λύση όταν δεν μπορούμε να πάρουμε τα, ε, η πρόσβαση, ε, αν δεν μπορούμε να πάρουμε πρόσβαση στα δεδομένα SWIFT. Εγώ νόμιζα ότι μέσω του SWIFT ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούμε να λάβουμε τα στοιχεία αυτά, τελεία και παύλα δεν έχω καταλάβει πολύ καλά και ελπίζω στην έκθεσή σας να αναφέρετε ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει μία ε, ε δίωδος άγγλισης δεδομένα από το SWIFT και παραπάνω. Επίσης μιλάτε για μια αξιολόγηση του συστήματος PNR σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά δεν απαντάτε το ερώτημα. Λέτε απλώς ότι επιτρέπει στο Υπουργείο το Αμερικανικό να κάνει καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου κλπ αλλά ποια, ποιες είναι οι αποδείξεις, ε, πού είναι οι αποδείξεις ε, και γιατί παρακολουθούμε τελικά τους ε, υπόπτους τρομοκρατίας. please, and please. Η κυρία Βερζιάτ, και σύντομα παρακαλώ. Ναι, θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο που ήρθε αμέσως εδώ μετά από την έκθεση που η Επιτροπή υιοθέτησε. Και όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν είχα το χρόνο να διαβάσω αυτά τα κείμενα έτσι στα πρόχειρα μόνο, στα πεταχτά και διάβασα στον τύπο αντιδράσεις και τα πρώτα που άκουσα συμφωνούν απόλυτα με τα σχόλια που απευθύναν, που έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοι σχετικά με την παρουσίαση, με τον τρόπο που μας προέρχονται τα πράγματα. Κύριε Επίτροπο, μας είπατε στο πρώτο μέρος για την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά της τρομοκρατίας και για την προστασία των πολιτών. Δεν είναι όμως ικανοποιητική αυτή η παρουσίαση. Την κολέρια Αέστ ε, να πω και εγώ ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικό για αυτή τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος με ποιες περιπτώσεις, ποιες περιπτώσεις αφορά το θέμα, αλλά γιατί, γιατί αποτελεσματικές. Θα πρέπει να ξέρουμε εμείς πώς ακριβώς η χρησιμοποιούμε διαδικασία που έχει να κάνει με την προστασία αυτών ε, είναι και αποτελεσματική κατά της τρομοκρατίας. Ε, δεν υπάρχει τίποτα, παραλαμβάνω, που να μας το αποδεικνύει. Στα κείμενα αυτά το λέτε και εσείς στην παρουσίασή σας για τη χρησιμότητα, για τη σημαντική αξία αυτών των συμφωνιών. Αλλά ποια είναι η αρχή, όχι η χρησιμότητα έτσι σκέτη, αλλά η απόλυτα απαραίτητη για να πετύχει κανείς στόχους και σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί αυτά παρακάμπτονται. Και ακόμα κάτι, άκουσα αρκετά και τις παρατηρήσεις για τη Europol, για την αρχή ελέγχου. Εκεί όμως δεν ισχύουν αυτά δυστυχώς. Ναι, εντάξει, εντάξει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρος, μην ανησυχείτε. Έτσι με μια κίνηση και δεν βασίζονται όλα αυτά πουθενά, κάτι τελευταίο και αναφέρθηκε νομίζω και αυτό λίγο πολύ. Τι μας λέτε ότι δεν έχουμε αντίθετες αποδείξεις. Ε, οτιδήποτε εμφανίστηκε στον τύπο από τον Ιούνιο δείχνει όμως ε, κάποιες υποψίες γενικές επί του θέματος εσείς ε, που βασίζεστε και να λέτε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη αντίθετη για το τι θίγεται και τελευταία να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις ε, Μπρεσ νομίζω ότι είναι από τα σημαντικά σημεία δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και το ίδιο ακριβώς είμαστε πάντα στην αφετηρία ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σοβαρές ανησυχίες ακούστηκαν. Αν θέλετε όμως να ακούσετε και τις απαντήσεις πρέπει να βιαστούμε λίγο. Κυρία Ρομέρο Λόπεζ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ναι, κυρία Μέλστραμ, αυτή τη δέσμη δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε αυτό το πρόσφατο κείμενο. Παντού σας ευχαριστούμε πραγματικά. Έχουμε αυτό το πρώτο μέρος γιατί όσοι έκαναν αυτή την αναθεώρηση δεν ε, έλαβαν υπόψη τους όλο αυτό το φαινόμενο το τελευταίο και είναι ε, όλα αυτά τα τελευταία, τα πολλά, ότι μετά πώς αποκαλύφθηκαν, δεν υπάρχει πια κλίμα εμπιστοσύνη ε, και εδώ θα πρέπει, ίσως θα έπρεπε να διακοπεί αυτό το PNR και θα πρέπει να καταλάβουν και οι Αμερικανοί και εκείνοι αυτά λένε ε, το τι συμβαίνει, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις υπηρεσίε κατασκοπίες. Νομίζω δεν υπάρχει πια κλίμα εμπιστοσύνη και από το ΕΛΚ επίσης που μίλησαν και είπαν ότι το PNR δεν θα πρέπει να ισχύει πια. Δεν είναι αυτή τη στιγμή για μια θεώρηση έτσι και για τη μελέτη αυτής της δέσμης. Δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη. Να δούμε πώς θα την αποκαταστήσουμε, τι θα κάνουμε για να αλλάξει η κατάσταση. Αυτά που συνέβησαν ήταν πριν ε, με την υπόθεση Snowden δεν άλλαξαν τα πράγματα. Όχι γιατί υπόθηκαν πράγματα που τα γνωρίζαμε. Αλλά κατάλαβαν οι Αμερικανοί ότι δεν μπορεί κανείς να καταδιώξει την τρομοκρατία χωρίς να σεβαστούν τις ανθρώπινες ελευθερίες δεν είναι στο τηλέφωνο της κυρίας Μέρκελ ο ε, και ούτε στη Βραζιλία. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει πια κλίμα εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να το αποκαταστήσουμε, να δούμε το πρόγραμμα πλαίσιο και για μια δικαστική αρρωγή. Και στα πλαίσια αυτό ίσως είναι διαφορετικό από ό,τι κάναμε, αλλά θα πρέπει Τώρα να εξετάσουμε αυτή τη δέσμη είναι σαν να είμαστε στον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο αιώνα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα τωρινά. Ευχαριστούμε. Βάιντερ Χάτερ. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι για το ότι ήρθατε τόσο γρήγορα, κυρία Επίτροπε, αλλά αυτό είναι το μόνο θετικό. Γιατί θεωρώ πως εδώ πέρα έχουμε μία διαδικασία όπου μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία. Εγώ θεωρώ πως δεν έχει κλείσει καθόλου αυτή η υπόθεση. Και δεν πρέπει να πούμε στους Αμερικάνους πως έχει τελειώσει χωρίς να συζητήσουν μαζί μας. Κάποιοι δεν είχαν δει τα έγγραφα το πρωί κάποιοι πιο νωρίς, εγώ το έλαβα ζεστό από το φωτοτυπικό, τώρα το διαβάζω και θεωρώ πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια συζήτηση και να διαβάσουμε νομίζω πριν από αυτήν τα έγγραφα. Αλλά δεν αρκεί να ρωτάμε το αν τηρήθηκε κάτι, αλλά χρειάζεται νομίζω μια πιο σοβαρή έρευνα και μέθοδος. Δεν έχει τελειώσει καθόλου αυτή η υπόθεση και το κεφάλαιο και νομίζω μπορούμε να το πούμε. Γιατί πρόκειται για παραβίαση της εμπιστοσύνης, δικαίως μιλήσατε για εμπιστοσύνη. Τους χρειαζόμαστε τους Αμερικανούς μας φίλους, αλλά αυτό το οποίο λείπει εδώ πέρα είναι η εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό διακινδυνεύεται εδώ πέρα με αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να σα ρωτήσω αν μπορείτε να αποκλείσετε πραγματικά την οικονομική κατασκοπία στο πλαίσιο των ε, υποκλοπών αυτών. Και με ενδιαφέρει και η ποσοτική διάσταση. Δεν μας είπα δηλαδή πόσους τρομοκράτες ή πώς τρομοκρατικές επιθέσεις εμποδίσατε. Και κάτι άλλο. Είναι ιδιαίτερος θετικό το ότι ε, ακούσαμε και τις απόψεις ε, και ακούσατε και τις απόψεις ε, των Αμερικανών βουλευτών, αλλά μην ξεχνάτε πως υπάρχουν και Ευρωπαίοι βουλευτές, στους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω η κυρία Κοράτσα Μπίλτ θέλει να πει κάτι σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Συνήθως δεν σχολιάζω πολύ σοβαρά και τεχνικά ζητήματα όταν δεν έχω διαβάσει την έκθεση και πραγματικά θαυμάζω ότι ε, οι συνάδελφοι έχουν τόσο λεπτομερή γνώση χωρί να έχουν διαβάσει τι εκθέσει. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τις Ηνωμένε Πολιτείε και να ρωτιέμαι αν αυτή είναι η σωστή στάση. Ακούσαμε αγανάκτηση, ε, απαράδεκτο και ότι ε, είναι λάθος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα κάνουμε, θα κηρύξουμε πόλεμο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι προτείνετε, θα είμαστε ο Νετανιάχου της Ευρώπης, δηλαδή Ακόμα και όταν ε, το ΙΠΑ και ε, η Ιράν ε, συνάπτουν μια φοβερή συμφωνία, ίσως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα μπροστά, να χρησιμοποιήσουμε το διάλογο. Σοφή, μιλήσαμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τους μιλάμε. Εμείς δεν είμαστε παγκόσμιο δικαστήριο, είμαστε σύμμαχοι με τις ΙΠΑ. και ξέρεις κάτι συγγνώμη, έχω το λόγο, Σοφή, είμαι με διακόπτης. Το θέμα δεν είναι το θέμα της ε, παρακολούθησης από την NSA που μας σοκάρει όλους. Μιλάμε για δύο συγκεκριμένες οδηγίες, ε, συμφωνίες. Συμφωνίες. Συμφωνία θα πει δύο εταίροι. Συζητούμε λοιπόν μαζί τους, κάνουμε διάλογο και δεν νομίζω ότι όλα αυτά που υπόθηκαν ή όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην, στην, στην επιστολή είναι ε, να μην αφορέ να μην έχουμε πια ε, συνεργασία με τις ΗΠΑ. Έχουμε αποφασίσει το αντίθετο, να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ και δεν λέω ότι είμαι ικανοποιημένη με αυτά που γίνονται, απλώς λέω δεν είμαστε δικαστήριο εδώ, προσπαθούμε να υπάρξει εμπιστοσύνη και με τους Ευρωπαίους πολίτες και με τους Αμερικανούς, ε, έχουμε παρόμοιους στόχους με τους συμμάχους μας, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμένα αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, όπως βλέπετε, κυρία Επίτροπε, είναι ένα πάρα πολύ ε, συναισθηματικά φορτισμένο ζήτημα ε, κάτι που δικαιολογεί βέβαια και το είδος των σχολείων που ακούσατε. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ε, με αυτό το θέμα της ε, παρακολούθησης NSA και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα την αποκαταστήσουμε, ακούγοντας ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε όλες αυτές τις απόψεις. Παρακαλώ λοιπόν, σας δίνω το λόγο, προσπαθήστε να απαντήσετε ή να σχολιάσετε όλα αυτά που ακούσατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, βεβαίως θα προσπαθήσω να απαντήσω Καταλαβαίνω ότι δεν διαβάσατε την έκθεση, Λυπάμαι πολύ, αλλά ε, Ήθελα να έρθω όσο το δυνατόν συντομότερα και α μην έχετε διαβάσει την έκθεση. Ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσει και αφού θα τα έχετε διαβάσει τα έγγραφα. Εμεί ευχαρίστω να έρθουμε κάθε φορά που μας μια, μια επιτροπή μα καλεί. Φυσικά η αποκάλυψη του τι συνέβη με την NSA έχει δημιουργήσει αγανάκτηση. Είμαστε εμεί ε, ε, αναστατωμένοι, όλοι είναι αναστατωμένοι ότι έχει γίνει κάτι το ανεξέλεγκτο αυτό που συμβαίνει πια στι ΗΠΑ ότι υπάρχει μαζική παρακολούθηση με τρόπο που είναι προφανώ παράνομο ε, υπό πολλέ έννοιε και φυσικά αυτό δεν είναι καλό και δεν είναι αποδεκτό και υπάρχουν πολλέ διαδικασίε που έχουν ξεκινήσει για να αποσαφινιστεί όλη η διαδικασία και να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Αυτό που εγώ προσπάθησα να κάνω είναι να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη συμφωνία, με το TFTP. Πριν από το Snowden είχαμε διαδικασίες που είχαν ήδη δρομολογηθεί, που είχαν υποσχεθεί ε, μία έκθεση για την προστιθέμενη αξία του TFTP, μία πρώτη έκθεση για το PNR, μία πρώτη αναθεώρηση για το πώς ε, ε, ε εκπληρώνουν τις εκ της συμφωνίας υποχρεώσεις τους. Έχουμε παραδείγματα για να το υποστηρίξουμε αυτό. Και επίσης να δούμε και τις διάφορες εναλλακτικέ επιλογές άντλησης δεδομένων από τις ευρωπαϊκές πηγές. Αυτό είναι ένα τμήμα της NSA, όχι το σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αγνοεί την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ζητήσατε αναστολή. Αν διαβάσετε τη συμφωνία TFTP, λέει ότι αν υπάρχει διαφωνία όσον αφορά την ερμηνεία ή την ε, πλήρωση των όρων ε, ε, της συμφωνίας, πρέπει να υπάρξει διαβούλευση και μετά από τη διαβούλευση αν δεν υπάρχει ε, συμφωνία, τότε μπορεί να, αναστολεί, να ανασταλεί συμφωνία. Ε, δεν μπορείτε απλώ να την αναστείλετε. Αυτό είναι παραβίαση τη συμφωνία. Αυτό που έκανα ήταν να αρχίσω τι διαβουλεύσει και δεν του πήρα τηλέφωνο να του πω Συγγνώμη, παρα, παρεύετε τη συμφωνία. Όχι. Α, πολύ ωραία, ευχαριστώ αφιέρωσα ώρες επί προσπαθώντας να ε, λύσω τα ζητήματα που θα δείτε και στα έγγραφα. Αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομία, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα, δεν μπορούμε να κάνουμε επιστημονικές έρευνες, μπορούμε μόνο ερωτήσεις και διάλογο να κάνουμε, γιατί αυτό κάνουμε με τους εταίρους μας και το κάναμε αυτό και σε μεγάλο βαθμό. Λάβαμε απαντήσεις, ε, λάβαμε ε, διευκρινήσεις, λάβαμε γραπτές διαβεβαιώσεις από το και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπήρξε παραβίαση. Μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι υπήρξε παραβίαση συμφωνία. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να τον το αποδείξουμε. Εκτό από κάποιου ισχυρισμού στον τύπο. Αλλά προφανώ αυτό δεν είναι παρκέ για να αποδείξουμε του ισχυρισμού αυτού και ότι υπήρξε παραβίαση. Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε, όπως βλέπετε και από την επιστολή του ε, κυρίου Κοέν, προσπαθούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη χωρίς να γίνει ένα διαπραγμάτευση της συμφωνίας, αλλά προσπαθούμε να δούμε πιο πολύ τις, ε, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι ε, αμερικανικές αρχές προστασίας δεδομένων, να έχουν μια καλύτερη ε, θεώρηση των πραγμάτων και να λάβουν υπόψη και τις δικές μας απαιτήσει ως προς την προστασία δεδομένων. Θα γίνει να θεώρηση την ε, ερχόμενη άνοιξη και ε, βεβαίως τότε θα έχουμε κάθε λόγο να το θέσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως έρχεται σε διαβουλεύσεις. Το Σώμα των Επιτρόπων σήμερα το πρωί αποφάσισε να κλείσει τις διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό, για αυτή την πτυχή Όσον αφορά την ποιότητα της ε, αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία στην συμφωνία TFTP. Πιστεύουμε ότι χρήζουν μεγαλύτερης βελτίωσης όσον αφορά την αποπροσωποποίηση των δεδομένων, περισσότερες πληροφορίες, δεδομένα στατιστικές, για να ε, κινηθούμε προς ένα σύστημα push ε, σε μεγαλύτερο βαθμό και αυτό βεβαίως ε, θα το συζητήσουμε μαζί σας και θα σας ε, αναφέρουμε ενδεχόμενη πρόοδο συστηματικά. Δεν έχουν όμως λύσει τα πάντα. Ε, εξακολουθούμε να ανησυχούμε και μας απασχολεί το τι έγινε ε, το τι έκανε η NSA ε, παρακολουθώντας και ιδιώτες και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο βέβαια σας ενδιαφέρει πολύ εσάς αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εντάξουμε και αυτή τη συμφωνία ο Μπρέλα, την ευρύτερη συμφωνία προς όφελος των πολιτών. Μπορείτε να ρωτήσετε και την Αντιπρόεδρο Ρέντιν όταν θα έρθει για περισσότερες λεπτομέρειες γιατί εκείνη γύρω των διαπραγματεύσεων αλλά εγώ ήμουν ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες και εκείνη την περασμένη εβδομάδα και συμφώνησαν με τους Αμερικάνους εταίρους να κάνουν ό,τι μπορούν πριν από το καλοκαίρι και ακούσατε ίσως και ότι ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι όταν μπορεί κανείς κάτι να κάνει δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει. Υπάρχουν λοιπόν πολλές συζητήσεις και ε, πολλά, ε, πολλές διαβουλεύσεις Όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η NSA δεν θα έχει ξανά τόσο σοβαρό αντίκτυπο στα ε, δεδομένα ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Όσον αφορά τώρα την άντληση των δεδομένων, τα, Swift, ε, τα δεδομένα SWIFT είναι ε, δεδομένα χίδιν. Δηλαδή δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο και λέει πείτε μου τι ξέρετε για τη Σοφή Ινετβέλτ. Οπότε πρέπει κανείς να δημιουργήσει ένα σύστημα άντλησης ε, δεδομένων σε ευρωπαϊκό ε, έδαφος. Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο βεβαίως, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι επιθυμητό, κατά πόσο είναι αναλογικό, κατά πόσο υπάρχουν σωστοί λόγοι να γίνει αυτό και να υπάρξει μια βάση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά το αφήνω σε εσά και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο για την ώρα δεν έχει δείξει καμία προθυμία και μετά την πρώτη ε, συζήτηση που κάναμε πριν από δύο χρόνια δεν υπήρξε κανένα συζητητής από την Επιτροπή σας και καμία σαφής ένδειξη από εσά για το πώς θα προχωρήσουμε. Τα αφήνω όμως σε εσά, μπορείτε να δείτε τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ιστότοπό τη, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να προτείνετε κάτι που η επόμενη Επιτροπή και η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία βέβαια θα το προχωρήσει. Τόσες πολλές ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε, πρέπει να με βοηθήσετε, μήπως ξέχασα κανέναν. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε λάβει όλες τις απαντήσεις. Ούτε και εμείς τις έχουμε λάβει όλες τις απαντήσεις που ζητήσαμε από τους Αμερικάνους στο ευρύτερο θέμα της NSA. Θα θέλαμε το Συμβούλιο να ήταν και λιγάκι πιο ε, συνεργάσιμο στις συζητήσεις του με τη ΣΥΠΑ, αλλά για την ώρα δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα πάντα ή συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη τίποτε έτσι έχουν τα πράγματα, θα προσπαθήσουμε να ε, παρακολουθούμε τα πράγματα, θα ε, πάρα πολύ ε, προσεκτικά και ευχαρίστως βέβαια να σας αναφέρουμε την πρόοδο. Ευχαρίστως να έρχομαι όποτε θέλετε. Πρόεδρος, ναι πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά την έκθεση, είναι σαφές, δεν είχαμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό και είναι χρήσιμο να, να συνεχίσουμε το διάλογο αυτό μετά από μερικές εβδομάδες αφού θα έχουμε διαβάσει τα έγγραφα και αφού βέβαια θα έχετε κι εσείς πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Και θα είμαστε και έτοιμοι για κάποιες συστάσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Γιατί είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να δούμε ξεχωριστά αυτό το θέμα από όλα τα υπόλοιπα. Συνδέονται μεταξύ τους και όλα αυτά συνδέονται και με την σχέση Ευρωπαϊκής ΥΠΑ. Αν μπορείτε κι εσείς, ε, μπορούμε και στο μέλλον να σας εγγράψουμε και πάλι στην ημερήσια διάταξή μας. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και σας ευχαριστώ και όλους εσάς συνάδελφοι που προσπαθήσατε να τηρήσετε τα χρονικά περιθώρια. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για το επόμενο θέμα που είναι η σύντομη ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Επιβολή του Νόμου αλλά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε παρά το ότι φάγαμε λίγο χρόνο από το θέμα αυτό.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 Okay. Uh, hello. Okay, I will give you the floor. <laughs> Sorry, I uh, we definitely uh, have to continue. Πρέπει να συνεχίσουμε. Λυπούμε πολύ παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο και επίμαχο θέμα να συζητήσουμε πιο πριν. Τώρα έχουμε ένα λιγότερο επίμαχο, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Επιβολή του Νόμου. Το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση του προγράμματος αυτού για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών ε, κυρίως στις μεθοριακές περιοχές και για την ενίσχυση της ε, κουλτούρας επιβολής του νόμου. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν υπάρχουν μόνο πολλές υπηρεσίες ευρωπαϊκές που εκπροσωπούνται σήμερα, ε, αλλά ότι είναι ε, και ακόμη περισσότερες που έχουν έρθει εδώ, που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε πολλούς ομιλητές για το απόγευμα. Η κυρία Ματιέ η οποία θα ήταν η εισηγήτρια. Ε, δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ για το θέμα αυτό του ΣΕΠΟΛ, κατά πόσο μπορεί η ΣΕΠΟΛ να είναι ανεξάρτητη από την ε, Europol, η οποία ΣΕΠΟΛ βέβαια πάρα πολύ επηρεάζεται από όλα αυτά τα προγράμματα κατάρτισης και θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση. Αλλά και εσείς ακούσατε τις απόψεις των διαφόρων ε, υπηρεσιών ε, και ήταν πολύ σαφής ε, η άποψη της ΛΥΜΠΕ κατά οποιασδήποτε συγχώνευσης μεταξύ, μεταξύ των δύο και το Συμβούλιο, 15 κράτη, 25 κράτη-μέλη είναι κατά της συγχώνευσης. Είναι σημαντικό αυτό το, αυτό το σχόλιο στο τμήμα της συζήτησης. Η κυρία Ματιού δεν είναι εδώ, Ο κύριος Πρίμπε τότε να λάβει το λόγο, επειδή ξέρω ότι χρειάζεται να φύγει νωρίτερα και μετά οι προσκεκλημένοι μας θα λάβουν το λόγο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί σύμφωνα με τα όσα γράφει το πρόγραμμά σας έπρεπε να έχω ήδη μιλήσει. Η Κομισιόν το Μάρτιο υιοθέτησε λοιπόν μια ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αστυνομικής εκπαίδευσης με στόχο να υπάρξει μια συντονισμένη ε, εκπαίδευση όλων των ε, αστυνομικών όλων των βαθμών, ειδικά σε ζητήματα διασυνοριακής αστυνόμευσης. Η αστυνόμευση πλέον έχει σαφή διεθνή διάσταση και η ευρωπαϊκή νοοτροπία των αστυνομικών είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη μιας κοινή αστυνομικής κουλτούρας. Ε, το, η πολιτική ενός συστήματος αστυνομικής εκπαίδευσης βασίζεται σε κάποιες δέσμες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η πρώτη δέσμη θα είναι βασικές γνώσεις για τα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη συνοριακή συνεργασία για όλους τους αστυνομικού. Δεύτερη δέσμη εις βάθος γνώση της καθημερινής συνεργασίας, ε, ειδικευμένα μαθήματα. Τρίτον, κοινά εκπαιδευτικά εργαλεία για αστυνομικέ αποστολές σε τρίτες χώρες και ε, εξαγωγή βέλτιστων πρακτικών σε τρίτες χώρες. Η ανακοίνωση κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των τεσσάρων δεσμών αυτών, με την έννοια ότι οι δέσμες 1 και 2 είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορούν να υποφεληθούν από το σύστημα αυτό όσον αφορά εργαλεία εκπαίδευσης, βέλτιστες πρακτικές, ενώ οι δέσμες 3 και 4 ε, είναι πιο στοχευμένες σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η ανακοίνωση παραδείγματος χάρη λέει πως στην τέταρτη θέσμη πως ε, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι βασικό κομμάτι του σχεδιασμού αποστολών σε τρίτες ε, χώρες και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση πριν την αποστολή ως προαπαιτούμενο για να αποσταλούν σε αποστολές τέτοιες αστυνομικοί. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ιδεώδης ευκαιρία για να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, αλλά και για να αναγνωρίσουμε τη σημασία του συντονισμού της εκπαίδευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση και να μην υπάρχουν, υπάρχει σπατάλη προσπαθειών και πόρων. Γι' αυτό ευχαριστούμε την ΣΕΠΟΛ που οργάνωσε την εκδήλωση αυτή και μάλιστα δεδομένων των προσπαθειών που έχουν αφιερωθεί σε αυτό. Νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη φάση της εφαρμογής. Η ανακοίνωση του Μαρτίου προβλέπει πως το ΣΕΠΟΛ θα είναι ε, η κινητήριος δύναμη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη Άλλε υπηρεσίε και ενδιαφέρομενου. Δεδομένων των περιορισμών στον προπολογισμό, είναι προφανέ πω κάποιε προθεσμίε που αναφέρονται στην ανακοίνωση δεν θα τηρηθούν, παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε για το ότι η ΣΕΠΟΛ αναγνωρίζεται ω κινητήριο δύναμη. Και τέλο θα ήθελα να προσθέσω Πώ έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε συζητήσει για το μέλλον τη ΣΕΠΟΛ, αλλά από τη δική μα την πλευρά τους τελευταίους μήνες μετανιώσαμε το ότι με την συζήτηση αυτή παραμελήσαμε λίγο να κοιτάξουμε την ουσία. Οπότε και πάλι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ευκαιρία να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Πάντα βεβαίως στο πνεύμα της επικουρικότητας, δηλαδή η βασική εκπαίδευση των αστυνομικών είναι βεβαίω υπόθεση των κρατών μελών ή περιφερειών αναλόγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούμε πω η εκπαίδευση των αστυνομικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε, τον λόγο έχει ο κύριο Σρέντερ από την ΣΕΠΟΛ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκπράσω την ευγνωμοσύνη μας για το ότι μας καλέσατε στην εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα να περιοριστώ σε τρία βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα επιτρέψατε μου να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του, της λειτουργίας της ΕΠΟΛ. Μετά θα κάνω κάποιες γενικές, παρουσία, κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το μέλλον και μετά βεβαίως να δούμε τα βασικά σημεία του συστήματος αστυνομικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, ξεκινώντας από την ΣΕΠΟΛ. Όπως ξέρετε, η ΣΕΠΟΛ βασίζεται σε ένα δίκτυο των σχολών της αστυνομίας στην Ευρώπη και αυτή είναι η δύναμή της. Δηλαδή, αφενός είμαστε συνεργασία με όλους αυτούς τους εταίρους, από την άλλη βεβαίως στηρίζουμε τους εταίρου μας εντός των κρατών για να προωθήσουν τις δραστηριότητες τους στο επίπεδο των κρατών μελών. Επίσης, αναζητούμε συνεργασία με άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ένωσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τη Europol, τη Frontex και τη Eurojust είχαμε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τελικά η βασική αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών ε, ενεπλάκη στην ε, όλη διαδικασία. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα υπάρχει επίσης καλή συνεργασία με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, τα αναγνωρίζουμε ως ε, κάτι το πολύ σημαντικό για όλες τις τυχές της εκπαίδευσης ε, των αστυνομικών. Βεβαίως έχουμε και συνεργασία με την ΕΑΣΑ, ΕΛΙΖΑ και τις λοιπές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα επιβολής του νόμου. Επίσης προσπαθούμε να κλείσουμε το κενό μεταξύ πολιτικής και πρακτικής ε, και βεβαίως ειδικά όσον αφορά την πολιτική. Ε, μπορεί να υπάρχει ένας ωραιότατος κανονισμός, αλλά θα πρέπει οι αστυνομικοί να μπορέσουν να εργαστούν με αυτό. Κάποιες βασικές πληροφορίες για το επιχειρησιακό μας μοντέλο ε, εμείς εμπλέκουμε όλους τους ενδιαφερομένους, δηλαδή τις ε, σχολές αστυνομίας, αλλά και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή μέχρι και την εφαρμογή ή όλες οι προτεραιότητες μας βασίζονται σε στρατηγική αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης και τώρα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις υπόλοιπες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γύρω στο 40% θα έλεγα της εκπαίδευσης αφιερώνεται σε αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες ε, εφαρμόζονται από τις σχολές και μέσα στις σχολές αστυνομίας των κρατών μελών. Έχουμε διάφορες επιλογές πέρα από τα κλασικά σεμινάρια. Ε, έχουμε και ηλεκτρονική διδασκαλία, έχουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής αστυνομικών, έχουμε επίσης ε, κοινή η ύλη και αναμένουμε επίσης να έχουμε πάνω από 7.000 συμμετέχοντες φέτος στις δραστηριότητές μας. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, στηρίζουμε τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες εκείνες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονία. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ΣΕΠΟΛ και το δίκτυό της παίζει ένα ρόλο κλειδί ήδη στην οικοδόμηση δυνατοτήτων των αστυνομιών στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε τώρα για μια κοινή αστυνομική κουλτούρα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο και θεωρούμε με τις δραστηριότητές μας πως το να έρθουν σε άμεση επαφή αστυνομική και να γνωριστούν και να μάθουν ένας από τον άλλον είναι κάτι το πολύτιμο όταν μιλάμε για την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει για το τι θα γίνει μετά τη Στοκχόλμη και εμείς προτείνουμε να υπάρχει σαφής ρόλος για την αστυνομική εκπαίδευση ως ε, ένα παράγοντος που θα υποστηρίξει τις άλλες δραστηριότητες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το ELTS, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή βάση. Επίσης, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε λιγότερου πόρους στο μέλλον και βεβαίως έτσι θα μπορέσουμε να εστιάσουμε και θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα στην ποιότητα. Για να δώσω κάποια παραδείγματα, θεωρούν πως για τη μελλοντική ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στην ποιότητα της δακταίας ύλης, πιστοποίηση παραδείγματο χάρη. Επίσης σκεφτόμαστε την ποιότητα των εκπαιδευτών και εκεί θα θέλαμε να έχουμε ένα σύστημα πιστοποίησης των εκπαιδευτών και την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την ποιότητα των συμμετεχόντων. Εκπαιδεύουμε τους σωστούς ανθρώπους. Ε, πρέπει να βελτιωθούμε και για το μέλλον αυτό, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι άσχημο νομίζω, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Επίσης πρέπει να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε με τους περιορισμένους πόρους μας. Τέλος, η ποιότητα του περιβάλλοντος μάθησης, ειδικά όταν μιλάμε για το διαδίκτυο, που θα είναι πιο σημαντικό στο μέλλον, πρέπει να επενδύσουμε και εκεί πέρα για τους αστυνομικούς. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα τώρα όπως αναφέρθηκε, η Κομισιόν ήδη παρήχε μια στήριξη για την ε, χαρτογράφηση του τι γίνεται γενικώ στην αγορά θα έλεγα της εκπαίδευσης αυτής και βεβαίως εκτιμούμε ιδιαίτερα τις ε, βασικές δομές ε, του συστήματος αυτού και θεωρούμε πως έχουμε μια ξεκάθαρη δομή ευθυνών για το εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν πως έτσι υπάρχει σεβασμός στην αρχή της επικουρικότητας και όταν μιλάμε για τον ρόλο της υπηρεσίας νομίζουμε πως ε, έχουμε νομίζω μεγαλύτερη συνεισφορά στη μετατροπή αλληλεπικαλύψεων σε συνέργειες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό με περιορισμένους πόρους. Και όταν μιλάμε για την εξωτερική διάσταση της αστυνόμευσης, θεωρούμε πως ο ρόλος των αστυνομικών αποστολών, προετοιμασίας αποστολών, πρέπει να είναι καλύτερος συντονισμός και των προσπαθειών, των προσπαθειών στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτύχουμε περισσότερα με περιορισμένους πόρους. Όπως είπα, θεωρούμε πως η ΣΕΠΟΛ είναι σε θέση να παίξει τον ρόλο αυτό... και βεβαίως αναμένουμε να συνεισφέρουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γορόβιο Λεόν από την Ισπανία, αν μπορείτε παρακαλώ εντός πέντε λεπτών, για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ξέρω ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στη ΘΕΠΟΛ που μου προσφέρει την ευκαιρία αυτή για να εκφράσω την άποψη των Κέντρων Εθνικής Εκπαίδευσης ε, για αυτό το θέμα, για την επιβολή του νόμου. Εδώ θα προσπαθήσω να σας προσφέρω μία άποψη να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό από το, μέσω του ισπανικού προτύπου το οποίο γνωρίζω. Τέσσερα-πέντε σημεία με αυτά θα ασχοληθώ από ισπανικής πλευράς ε, τι γίνεται με την ασφάλεια που εξαρτάται από το κράτος, ε, ποια είναι η εκπαίδευση στην Guardia Civil και στην Εθνική Αστυνομία, αυτά είναι τα δύο κύρια, όπως επίσης ε, να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν ε, για τις βάσεις ε, για αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης ε, σε εθνικά κέντρα των κρατών μελών. Αυτό είναι το αστυνομικό πρότυπο, το ισπανικό, αλλά με ένα ειδικό χαρακτήρα. Υπάρχουν διάφορες αστυνομίες, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν Πολλές ομοιότητες επίσης με αστυνομικά σώματα στην Ευρώπη. 5,2 η αναλογία με τον πληθυσμό και έχουμε 155.000 αστυνομικούς στο σύνολό τους. Έχουμε την Guardia Civil και την ε, αστυνομία, την εθνική και με κατάλληλους μηχανισμούς ε, ε, συνεργασίας πραγματικής ανάμεσα σε όλα τα αστυνομικά σώματα. Αυτά που σας είπα πριν, 155.000 και κάτι αστυνομικούς και που είναι ανάμεσα στην Εθνική Αστυνομία και στην Guardia Civil για να δείτε ποιους αφορά αυτή η κατάρτιση. Έχει να κάνει με το σύνολο των αστυνομικών στη χώρα. Σε ποιες συνταγματικές αρχές βασίζεται το, ευρωπαϊκό, το πρόγραμμα αυτό κατάρτισης είναι μια διαφάνεια βέβαια και από θεσμικής πλευράς ορισμένα στοιχεία που εμφανίζονται στην ειδική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και έρευνας για να δείτε τις γενικές γραμμές από πού προέρχονται για αυτή την ε, αστρομική κατάρτιση είναι από το Συμβούλιο Υπουργών και μετά από το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Και, και με κατάλληλα προγράμματα, με και υπάρχουν οι επικεφαλής κατάρτισης στην αστυνομία και στην Guardia Civil. Είναι σωμετωμένα όλα αυτά στο γενικό σύστημα κατάρτισης με δική τους δομή. Και βλέπουμε τα διάφορα τμήματα που είναι οι ακαδημίες, οι επιχειρησιακές μονάδες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθηγητές, Φοιτητέ και μετά οι επιτροπές που κατευθύνουν τις καταρτήσεις όπως πρέπει ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Μόνο τρεις διαφάνειες για την όλη δομή στην Guardia Civil, επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση και υψηλού επίπεδου σπουδών και αυτή η διαφάνεια δείχνει παντού τη συνεχιαρχική εκπαίδευση, μετά η εξειδίκευση και μετά η ανώτατη εκπαίδευση. Θα ήθελα να σας πω ότι το σύστημα κατάρτισης ε, είναι απόλυτα ενσωματωμένα τα προγράμματα αυτά στη πλαίσια και τα ευρωπαϊκά σύμφωνα με τις αρχές που ισχύουν στο ε, σχέδιο της Μπολόνια και ένας ε, έχει ας πούμε ένας ε, υπολοχαγός ο οποίος ε, έχει διδάσκεται και τελικά έχει ένα ανώτατο δίπλωμα ουσιαστικά. Το ίδιο και στην αστυνομία έχουμε μια αρχική κατάρτιση, μετά ε, ανεβαίνει στους βαθμούς και μετά μια εξειδίκευση και ανώτατες σπουδές. και υπάρχουν διάφορα μέσα πρόσβασης, βλέπετε αυτές τις κατηγορίες σε αυτό το σχεδιάγραμμα. Και να σας πω ότι και στην αστυνομία εκεί έχουμε ε, ε, προσαρμόσει με έναν επιθεωρητή τελικά που έχει ένα μάστερ πανεπιστημιακό σύμφωνα με τα κριτήρια της Μπολόνια Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει ένα πασημιακό δίπλωμα και μετά από δύο χρόνια με το μάστερ έχει ακριβώς σε επίπεδο μάστερ που προσφέρεται από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Θα να σας πω ότι τα κέντρα αστυνομικής κατάρτισης ε, εκεί, στα κρατημέλη, ε, όλα αυτά υπάρχουν οι προϋποθέσεις των κέντρων αριστείας ε, και έχουν παρόμοια διαπιστευτήρια μέσω πιστοποίησεων ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ISO κλπ. Είτε το DFP. Και Επίσης και η Ευρωπόλ ελέγχει τα πράγματα και αυτό προσφέρει εγγύησεις κατάλληλες. Μετά από όλα σας είπα, για να δούμε, για να αναρωτηθούμε ακριβώς Υπάρχουν οι βάσεις για μια πραγματική επιβολή έτσι στα κράτη-μέλη. Ναι, υπάρχουν οι βάσεις γιατί είναι προσαρμοσμένα τα συστήματα με την ανώτατη στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή και σύμφωνα με τα κριτήρια της Μπολόνια και μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και ταυτόχρονα στην οργή κατάρτιση όπως και στην εξειδίκευση Εύκολο είναι να υπάρξουν να ισχύσουν οι προϋποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης όπως απαιτούνται από τα κρατημέλη τα στοιχεία αυτά. Και ακόμα κάτι για να δούμε πώς έχει όλη η εφαρμογή αυτού του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος Κατάρτισης εδώ εκεί που ανήκει σε ΠΟΛ. Σαν τμήμα θα πρέπει να έχουμε όμως και τους απαραίτητους πόρους και την υποστήριξη σε κάθε επίπεδο και ε, με την ε, στήριξη επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπολείπτων ε, φορέων σε ευρωπαϊκό πάντα επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρεις ακόμη παρουσιάσεις θα ακούσουμε. επειδή ο κύριος Πρίμπεμους θα πρέπει να φύγει, αν έχετε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι, να ζητήσω από τους επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ, στο Προεδρείο. Κύριε Μπρόνς, παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Πρίμπε. Ναι, θα προσπαθήσω. Έχω ξεχωριστά ερωτήματα για κάθε ομιλητή. ποιος ε, είναι το αντικείμενο της ε, κατάρτισης, ε, αστυνομία των κρατών μελών, η ΣΕΠΟΛ, μιλάμε για μεθοριακούς, μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, ανθρώπους που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, τι ακριβώς αφορά η κατάρτιση, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, τεχνικές εντοπισμού ή μιλάμε για... Ε, για ουσιαστικό δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εμείς ε, ε ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα της συγχώνευσης ή γιατί η Κομισιόν ήθελε να εξοικονομήσει κάποια λεφτά. Το ΔΕ Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου επέτρεψε πρόσφατα την εκπαίδευση αστυνομικών. Και μιλάμε για ένα 40% του προπολογισμού του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και ο κύριος Ρέντερ ανέφερε πως πως ήταν δύσκολο ακόμα και να καταγράψει ποιος εκπαιδεύει ποιον. Και παράλληλα με αυτή την καταγραφή υπάρχει μια άλλη διαδικασία σε πολλές ε, σχολές αστυνομία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ακριβώς τι κάνει η Κομισιόν. Thank you very much, Mr. Thank you for helping me. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με βοηθήσατε. όπως είπε ο κ. Μπρόνς, οπωσδήποτε κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Όλα αυτά τα οποία είπατε είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν καθοριστεί. Η βασική ιδέα του συστήματος είναι να εκπαιδεύσουμε αστυνομικού. Mm. των κρατών μελών που στέλνουμε στην Ευρωπόλ. Κατηγορίες τώρα εκπαίδευσης αστυνομικής. Αυτό σχετίζεται με τις τέσσερις δέσμες που ανέφερα. Οπωσδήποτε δεν έχουμε στόχο να περιορίσουμε το σύστημα αυτό μόνο σε αστυνομικού που κάνουν διασυνοριακές επιχειρήσεις. Ε, αυτή είναι μία προτεραιότητα. Γνωρίζοντας πως όλο και περισσότεροι αστυνομικοί βρίσκονται σε καταστάσεις όπου πλέον ε, εργάζονται διασυνοριακά, είτε μιλάμε για τα βελγικά σύνορα, είτε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. αλλά δεν τίθεται ζήτημα μείωσης ε, της εκπαίδευσης ε, και περιορισμού της ε, σε μεθόδους ανείχνευσης. Προσπάθησα να εξηγήσω πως η πρώτη δέσμη είναι να δουν το κομμάτι της δουλειά τους που αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία. Και να εκμεταλλευτεί αυτά τα οποία προσφέρει η Γεροπόλ. Όπως ξέρετε, συζητάμε αυτή τη στιγμή για τη Γιούπολ και βλέπουμε πως η ενημέρωση εθνικών αστυνομιών για το τι μπορεί να κάνει η Europol διαφέρει. Αναχώρα και περιφέρεια. Οπότε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε εντάσσονται σε αυτό το σύστημα. Δεν έχουμε αυτό σημείο να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και το άλλο, που εξάλλου δεν πρέπει να το πει η Κομισιόν. Απλά βρήκαμε τέσσερις τομείς όπου πραγματικά υπάρχει μια διάσταση πέρα από την εθνική. Για το ερώτημά σας τώρα. Δεν το ήξερα αυτό το οποίο λέτε, αλλά μου λένε εδώ πέρα πως είναι ένα διετές έργο, αλλά δεν μοιάζει να έχει σχέση με εκπαίδευση. Βεβαίως θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αντιφατικό να προωθήσουμε αυτό το σχέδιο αστυνομικής εκπαίδευσης όταν μιλάμε για περικοπές, αλλά γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να βρούμε λύσεις για να οργανωθούμε. Αλλά να επαναλάβω αυτό το οποίο υπάρχει κά, είναι σημαντικό να υπάρχει μια αντίληψη της ε, πολιτικής αυτής και μετά βεβαίως να βρούμε το πώς καλύτερα θα την εξυπηρετήσουμε. Εξάλλου μετά από όλες τις συζητήσεις που έχουμε για τόσα θέματα στον τομέα αυτών, νομίζω πως είναι αρκετά ελκυστικό ευρωπαϊκό έργο σε έναν τομέα όπου η εκπαίδευση και η νεοτροπία των αστυνομικών είναι εθνική ακόμα, χωρίς να αποτελεί αυτό σημείο κριτικής, αλλά η εγκληματικότητα είναι πλέον διασυνοριακή. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε βέβαια ότι η κατάρτιση των, ε, ε, των οργάνων επιβολής του νόμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν ε, για την παρουσία σας εδώ. Αν έχετε κάποιο χρόνο στο μέλλον, ευχαρίστως να συνεχίσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Uh, first, uh, thank you for coming here. Uh, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας εδώ και να ζητήσω από τον κύριο Φάρνχελμ, Φάρνχελμ από τη Frontex να πάρει το λόγο. Πέντε λεπτά παρακαλώ έχετε στη διάθεσή σας για να έχουμε και συζήτηση μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το πλαίσιο ε, προδιαγραφών για τους ε, συνοριοφύλακες και πώς συνδέεται με το όλο πρόγραμμα κατάρτισης. Η Frontex έχει ένα πάρα πολύ, μια πολύ συγκεκριμένη εντολή για κατάρτιση των συνοριοφυλάκων, κάτι το οποίο αναφερόταν ήδη ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε ότι έλεγε, λέγαμε δηλαδή ότι τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να ε, φυλάσσονται από ε, ιδιαίτερως εξειδικευμένους ε, φύλακες. Η Frontex πρέπει να συνεπικουρεί τα κράτη-μέλη στην εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών με την δημιουργία κοινών προδιαγραφών κατάρτισης. Βάσει λοιπόν των συμπερασμάτων αυτών ε, και του προγράμματος Στοκχόλμης και της, στρατηγικής, ε, της προγράμματος εσωτερικής στρατηγικής αλλά και βάσει της διαδικασίας της Μπολόνιας και της ε, Κόπενχάγης, δεδομένου ότι η Μπολόνια αφορά την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Όλα αυτά επικεντρώνονται στην εναρμόνιση, στις κοινέ προδιαγραφές, τη διαφάνεια, την κινητικότητα και την εξασφάλιση ποιότητας. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, το πλαίσιο ευρωπαϊκών προσόντων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ε, και η διαβίου εκμάθηση είναι το βασικό μέσο για την επίτευξη της κινητικότητας και της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμφωνήσαμε το 2008 και δημιουργεί κοινά, κοινές προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών διαβίου εκμάθησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος ε, έχει ή τουλάχιστον είναι στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εθνικού πλαισίου ε, ανάπτυξης προδιαγραφών ε, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχει εθνικά στοιχεία και πολιτικές, ε, είναι τέλος πάντων μια μεταγραφή όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων κατάρτισης και προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο, γιατί όλα αυτά εντάσσονται και συγκρίνονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν ήδη πολυάριθμα τέτοιου είδους προγράμματα ε, στο επιχειρηματικό δίκαιο και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά για τη φύλαξη των συνόρων ειδικότερα ε, η διαδικασία υπόκειται στην κατάρτιση οργάνων επιβολής του νόμου. Παρά το ότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφορετικών φορέων ε, φύλαξης συνόρων, ε, το SQF ε, ασχολείται όλος ιδιαίτερος με τους ε, σύνοριοφύλακες, επικεντρώνεται ειδικότερα στα καθήκοντα αυτά. Αναφέρεται συγκεκριμένα στα καθήκοντα αυτά, τα περιγράφει επακριβώς και τα ξεχωρίζει από άλλες από άλλες, άλλες, άλλες κατηγορίες καθηκόντων η Frontex πρέπει να επιβεβαιώνει αλλά και να διευκρινίζει περισσότερο το πλαίσιο αυτής της κατάρτισης. Το SQF είναι ένα σύνολο κοινών προδιαγραφών, συνοριοφυλάκων και ε, αποτελεί ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους συνοριοφύλακες. Ε, σημαίνει πολύ καλή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ε, Προγράμματος Κατάρτισης βάσει της εντολής κάθε υπηρεσίας. Ε, τα SQF για ε, κάθε ε, για τους συνοριοφύλακες μπορεί να συμπληρωθούν με την κατάρτιση άλλων τομέων, όπως για παράδειγμα των τελωνίων, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βολόνιας και της Κοπενχάγης και σε συνεργασία βέβαια με τις εθνικές αρχές. Αυτό σημαίνει συντονισμένη προσέγγιση βέβαια για τον τομέα αυτό ε, συμμετέχει στην καλύτερη ανάπτυξη της ε, κατάρτισης ε, και την αποφυγή της διπλής δουλειάς Το πλαίσιο είναι περίπου ίδιο ε, για τους συνοριοφύλακες όπως είναι και για τις ε, δυνάμεις επιβολής του νόμου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεκινήσει με ε, συγκεκριμένη χαρτογράφηση των καθηκόντων, των διαφόρων ε, εργασιών και στη συνέχεια να περάσει ε, στην πιστοποίηση. Η συγκριτησιμότητα είναι τεράστια σημασίας. Επειδή η Frontex ε, εφαρμόζει το πλαίσιο κατάρτισης και επίσης έχει αρχίσει τη μετάφραση του SQF και ε, την ε, ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνοριοφύλακες, ε, το πρόγραμμα κατάρτισης για την επιβολή των νόμων του νόμου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συνοριοφύλακες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Frontex έχει συνεισφέρει λοιπόν σημαντικά στην εφαρμογή ε, του ε, προγράμματος κατάρτισης ε, επιβολής του νόμου με ένα πλαίσιο ειδικά για τους συνοριοφύλακες και επίσης προσπαθεί να αυξήσει τη γνώση της για τη μεθοδολογία του προγράμματος SQF βλέποντας τι συμβαίνει στους υπόλοιπους τομείς. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι ειδικότερα ο τομέας των συνοριοφυλάκων και η κατάρτισή του συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε τη δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα να ζητήσω τώρα από την κυρία Ιγγιγκορ να πάρει το λόγο από τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ε, από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εμείς βεβαίως είμαστε ενσωματωμένοι στο, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και προσπαθούμε να φέρουμε την διάσταση ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να δώσουν στοιχεία και να βοηθήσουν τις υπηρεσίες δικαιοσύνης εσωτερικών στο να έχουν κάποιες επιχειρησιακές απαντήσεις. Ε, Παραδείγματο χάρη, να μιλάμε για την καταπολέμηση εμπορίου ανθρωπίνων όντων, μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τις υπηρεσίες δικαιοσύνης και εσωτερικών, τότε εμείς σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες προσπαθούμε να ε, φέρουμε και την προοπτική του θύματος. Για να σας δώσω μια ιδέα της συνεργασίας. Βεβαίω, προσπαθούμε να έχουμε και μια ανάλυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη δουλειά των υπηρεσιών αυτών. Είναι θετικότατο λοιπόν το ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν θεωρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα ένα βασικό κομμάτι γνώσης ε, Πρέπει να δούμε δηλαδή την αστυνόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να φαίνεται αυτό και στην εκπαίδευση. Οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν τη γνώση και τα μέσα που θα τους δώσουν δυνατότητα να είναι επαγγελματίες. Τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνέλεξε πολλά στοιχεία που αφορούν την αστυνόμευση και την εκπαίδευση στην αστυνόμευση. Εξαιρετούμε τους ανθρώπους ε, για τις διακρίσεις, τον αντισημιτισμών ε, εγκλήματα μίσους, ε, π.χ. εις βάρος ε, ΛΟΑΔΑ. Τα βασικά ευρήματα των ερευνών είναι πως υπάρχει θυματοποίηση και δεν αναφέρονται αυτά στην αστυνομία. Σημαντικό εύρημα. Πρέπει να έχουμε κατά νου στην, κατά την εκπαίδευση των αστυνομικών. Ένα από τα πράγματα που εξηγείται Ε, όταν μας λένε ότι δεν πάει ο κόσμος στην αστυνομία είναι το ότι δεν, δεν πιστεύουν ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει κάτι. Και υπάρχει ο φως διακριτικής μεταχείρισης από την αστυνομία. Δεν θέλω να αναφερθώ στην προηγούμενη συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, αλλά νομίζω πως είναι και βασικό μήνυμα για την αστυνομία, γιατί η οικοδόμηση εμπιστοσύνη με την αστυνομία με όλα τα μέρη της κοινωνίας εξίσου. Γι' αυτό είναι θεμελιώδες. Και η εκπαίδευση λοιπόν έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάνκε τώρα από τη Europol έχει το λόγο για πέντε λεπτά ακόμα. Uh, ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να με εδώ σήμερα. Ε, ευχαριστώ ε, πάρα πολύ τη Frontex και την Επιτροπή σας. Θα ήθελα να τονίσω επί τη ευκαιρία την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με, CIPOL, με τη ΣΥΠΟΛ, ΣΕΠΟΛ στα ζητήματα κατάρτισης. Να σας εξηγήσω τι κάνουμε στη Europol Στη Europol ε, λαμβάνουμε συχνά αιτήματα από τα κράτη-μέλη να υπάρξει επιχειρησιακή κατάρκιστηση για τις τεχνικές επιβολής του νόμου ή για την εγκληματολογική ανάλυση. Επίσης έχουμε ασκούμενους στην Europol από τα κράτη-μέλη. Οπότε λοιπόν ε, μας χαροποίησε ιδιαίτερα όταν μας ε, ζήτησε η ε, Frontex ε, να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης για την Επιβολή του Νέου. Μου. Ελπίζουμε να έχουμε μια διαρθωμένη προσέγγιση ώστε η κατάρτιση να είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα κατάρτισης θα συμβάλλει σημαντικά στην ανταλλαγή γνώσεων και στη σύγκριση προδιαγραφών στον τομέα. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα βοηθήσει στην δημιουργία δεξιοτήτων και γνώσεων ε, που χρειάζονται ε, οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το διασυνοριακό έγκλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΣΕΠΟΛ πρέπει να παίξει σημαντικό και κρίσιμο ρόλο ε, στο πρόγραμμα ε, κατάρτισης. Όπως είπε και ο κύριος Σρόντερ, η ΣΕΠΟΛ έχει άμεση πρόσβαση στην κατάρτιση και στις γνώσεις ε, ε, μέσω των εθνικών αστυνομικών ακαδημιών και τα τελευταία χρόνια η Europol και η ΣΕΠΟΛ συνεργάζονται αποτελεσματικά. Γίνονται μαθήματα στο πλαίσιο της ΣΕΠΟΛ. Έχουμε ήδη αναπτύξει πολλά προγράμματα μαθημάτων, ειδικότερα στον τομέα της εγκληματολογικής ανάλυσης, αλλά και για συγκεκριμένους ε, τομείς, όπως στην περίπτωση των εγκλημάτων στο κυβερνοχώρο. Η συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και προδιαγραφών. Για την ώρα, για παράδειγμα, έχουμε προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Εκπαιδεύουμε αυτούς που πρέπει να εκπαιδεύσουν ε, αστυνομικούς στις χώρες τους, η ε, ηλεκτρονική εκμάθηση, ανάπτυξη προγραμμάτων και λοιπόν. Επίσης στο μέλλον ευχαρίστως ε, θα συμμετέχουμε με διαλέξεις, με κάθε δυνατότητα που υπάρχει στο πλαίσιο του επαγγελματικού δικτύου για να μπορέσει να στεφθεί με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης θα είναι αποτελεσματικές ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για μια κουλτούρα ε, επιβολής του νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Έχουμε μία σαφέστερη εικόνα τώρα για το πρόγραμμα κατάρτισης στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν Υπάρχουν ακόμη ευρωβουλευτές για να θέσουν ερωτήματα. Ναι, δεν είναι και πολλοί οι συνάδελφοι που είναι παρόντες. Έχω εγώ ένα ερώτημα προς τον κύριο Βέρνχελμ. Συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας, λέει η Πρόεδρος. είχαμε μία συνάντηση για την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα ασύλου ε, μεταναστών που φτάνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι βέβαιη ότι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση τώρα. Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες γιατί η Frontex αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτές αυτές τις ανεξάρτησες ε, καταγγελίες λέγοντας ότι υπάρχει ένας ε, ειδικό υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Ίσως όμως θα έπρεπε να το συζητήσουμε και εμείς εδώ κάποια χρονική στιγμή. Ίσως θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε αυτή την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Συγγνώμη, λέει ο κύριος Φάνιχεμ, αλλά νομίζω ότι είμαι ο λάθος άνθρωπος ε, για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Το γνωρίζω, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο για να απαντήσει. Εντάξει, λέει η πρόεδρος. Η κυρία Ιγγινγκερ θα πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Απλώς ως υποσημείωση, εγώ είμαι τμήμα του Συμβουλευτικού Φόρουμ ε, που βασίστηκε στη δική σας πρωτοβουλία και που έχει συμπεριληφθεί στον εσωτερικό κανονισμό της Frontex για ε, την καθοδήγηση των κρατών μελών από τη Frontex σε τέτοιου είδους ζητήματα, είτε διαρθρωτικά, ε, είτε από συστηματικής απόψεως ε, για τις ε, μεμονωμένες καταγγελίες. Αποκινούμε διεθνείς ε, οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών συνεργαζόμαστε για να υπάρξει ένας μηχανισμός παρακολούθησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και ενδεχόμενες μεμονωμένες καταγγελίες που λαμβάνουν χώρα σε κοινέ επιχειρήσεις της Frontex. Σας το λέω αυτό ενημερωτικά απλώς. Ίσως ε, στην ευρύτερη συζήτηση για τον Ευρωπαίο Διαμισολαγητή να μην μας διαφεύγει το δυναμικό ε, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο ευρύτερων ε, καταγγελιών, ε, σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω όμως και ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο κύριος Μπρόντς. Uh, uh, down to those which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 υπάρχει στην εκπαίδευσή μας, στη Frontex. Ανεξαρτήτως του που εστιάζουμε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα υπάρχει. Μόλις ανέφερα τα προσόντα των συνοριοφυλάκων, τα θεμελιώδη δικαιώματα επίσης είναι μέρος του πλαισίου αυτού και όπως είπαμε έχουμε και αστυο, αστυνομικό θεμελιωδών δικαιωμάτων που διασφαλίζει το ότι γνωρίζουμε αυτά τα ζητήματα και παρά το ότι πάντα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας ε, και σεβασμού των δικαιωμάτων νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στο πρώτο και στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ που μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Νομίζω θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή.